då tänker jag... start the meeting, um, take your seat. Καλημέρα, ξεκινούμε τη συνεδρίαση. Πάρτε τη θέση σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Είναι πολύ σύντομη, μισή ημέρα γιατί ακυρώθηκε η απογευματινή συνεδρίαση. Λοιπόν, πρώτο σημείο, έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για ε, τροποποίηση, οπότε θεωρείται εγκεκριμένη. Θα περάσω τώρα στις ε, του Προέδρου στο επόμενο σημείο. Σήμερα... Δεν ξέρω πώς το λένε καν στα σουηδικά αυτό, το γλωσσικό καθεστώς, language regime what you say in, in, men, eh, eh, de eh, språk som finns... Ποιες είναι λοιπόν οι διαθέσιμες γλώσσες για τη διερμηνία. Det som normalt brukar vara är att danska... Είναι η συνήθις, ε, δανέζικα, εστονικά, τσεχικά και σλοβαϊκά δεν έχουμε, δυστυχώς. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες υπάρχουν. Υπάρχουν τώρα θέμα των διαθεσμικών μηχανισμών για την ισότητα των δύο φύλων. Στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει τελικά η σχετική εκδήλωση, αναβλήθηκε και στις 8 Δεκεμβρίου στην επόμενη συνεδρίασή μας ε, θα ακούσουμε από, τη, από το ε, Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα πληθυσμιακά ζητήματα μία ε, παρουσίαση. Έχουμε την έγκριση των ε, πρακτικών της σύσκεψης των συντονιστών. Έχει μοιραστεί έχουν μοιραστεί τα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να επισυνάψουμε τα πρακτικά της συνεδρία των συντονιστών στα πρακτικά της συνεδρίασή μα. Σημείο 4. Έγκριση των ε, πρακτικών συνεδρίασης της 3 η Σεπτεμβρίου. επισυνάπτεται και αυτά, ε, επισυνάπτονται και αυτά τα πρακτικά. Και πάμε στο επόμενο σημείο. Θα διεξαχθεί συζήτηση με εκπρόσωπο της μονάδας του ΙΕ για τις γυναίκες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας επισκέπτεστε. Η μονάδα του ΙΕ για τις γυναίκες είναι σχετικά νέος θεσμός. Όμως τα θέματα των οποίων επιλαμβάνεται απασχολούν εδώ και πάρα πολύ καιρό τον ΟΗΕ και συνεργαζόμαστε αγαστά με την μονάδα αυτή, από πλευρά δηλαδή της Επιτροπής μας και επιχαίρουμε ιδιαίτερος για τη συνεργασία αυτή Ε, θα ε, ήταν σκόπιμο ίσως να ακούσουμε μία παρουσίαση και μετά να αρχίσει η συζήτηση. Υπάρχει και το θέμα της Διεθνούς ε, ημέρας του ΟΗΕ για τα κορίτσια, νερά κορίτσια και στις 25 Νοεμβρίου είναι η μέρα του ΟΗΕ κατά της βίας, κατά των γυναικών και αργότερα σήμερα θα γίνει μία ψηφοφορία για διάφορες σχετικές προφορικές ερωτήσεις που θέλουμε να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα για να διαπιστώσουμε ποιο τρόπο θα ήταν σκοπιμότερο να προετοιμαστούμε για την επίσκεψη στο CSV το Μάρτιο του 2013 θα γίνει μια αποστολή στη Νέα Υόρκη και στον ΟΗΕ γιατί θα παραστούμε σε μία εκδήλωση για την κατάργηση και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα πραγματευτεί ο ΙΕ το θέμα και κυρίως που θα συνεργαστούμε, διότι όντως μπορούμε να συμβάλλουμε ενεργά. Η κυρία Μανιούν, που είναι η ειδική εντεταλμένη του ΟΗΕ για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, μας ε, είπε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να συναυθεί νέα διεθνή σύμβαση για αυτό το θέμα. Με αυτή λοιπόν την ε, συνοπτική παρουσίαση καλωσορίζω την κυρία Ντάγμα Χουνίκερ που είναι επικεφαλής της μονάδας ε, στο γραφείο των Βρυξελών. Θα σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μετά θα ακούσουμε τις ε, ερωτήσεις ε, των βουλευτών. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Μιχαήλα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Χάρηκα πολύ όταν πήραμε την πρόσκληση να έρθουμε σήμερα και να μιλήσουμε κυρίως για τη δουλειά για τις γυναίκες εδώ στις Βρυξέλλες και τι θα κάνουμε ως ε, οργάνωση για την 25η Νοεμβρίου, όπως είπε και ο Μάικλ, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της βίας στις γυναίκες. Μετά θα προετοιμάσουμε το θέμα της θέσης των γυναικών, το, Μάρτιο θα γίνει αυτό, και μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Γυναικών του Κοινοβουλίου θα έρθει επίσης. Επίσης, ε, τι έγινε στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρα των κοριτσιών που για πρώτη φορά γιορτάστηκε φέτος. Πρώτο θέμα. Το έργο των UN Women στις Βρυξέλλες. Υπάρχουμε εδώ και δύο χρόνια. Τα κεντρικά μας είναι στη Νέα Υόρκη και ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο Μίχαελ Μπάσελε, ο πρώην πρόεδρος της Χιλής. Και όταν ε, ενσωματώθηκαν γυναίκα. Η πρώην πρόεδρος της Χιλής λοιπόν. Ε, εμείς ε, συνδυάσαμε την επιχειρησιακή μας δουλειά και αυτό αύξησε την δύναμη που έχουμε. Και τα θέματά μας αφορούν και τα επιχειρησιακά θέματα και τα κανονιστικά. Εις ό,τι αφορά το γραφείο μας εδώ, εμείς έχουμε ένα μικρό, είμαστε ένα μικρό γραφείο σύνδεσμος ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι από τα λίγα γραφεία συνδέσμων που έχουν οι γυναίκες, αλλά η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σημασία. Η εντολή μας είναι να συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και εκτιμούμε και τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας αλλά και με τις άλλες Επιτροπές του Κοινοβουλίου. Με την Κομισιόν επίσης συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με το Συμβούλιο. Δεν δουλεύουμε τόσο στενά με τα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά αν χρειαστεί το κάνουμε ευχαρίστως. Και τι κάνουμε. Κυρίως δουλεύουμε πάνω σε δυνατότητες πολιτικού διαλόγου, κοινή διαμεσολάβησης, κοινό προγραμματισμό και γι' αυτό χαιρόμαστε διότι τον Απρίλιο φέτος, όπως ξέρετε ίσως, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την, ε, το UN Women για να ενισχύσουμε τη συνεργασία, τις ε, συμπράξεις και η ομάδα εργασίας για να καταρτιστεί το μνημόνιο συνεργασίας συνίστατο από μια ποικιλία εμπλεκομένων από την Κομισιόν και επίσης αναθεωρήθηκε και εξετάστηκε και από τα κράτη-μέλη. Αυτό το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα γιατί ήταν μια ολιστική προσέγγιση. Ποιος είναι ο σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει από την Κελέδη Άστον, την Μισελ Μπασλέ, από τις γυναίκες, είναι να δούμε πώς θα συνεργαστούμε πιο στενά για την κοινή διαμεσολάβηση, τον πολιτικό διάλογο και τον κοινό προγραμματισμό. Και εκεί έχουμε κάποια επιτεύγματα να αναφέρουμε. Μόλις υπογράψαμε ένα μεγάλο καινούριο πρόγραμμα για την ενίσχυση των γυναικών πολιτικά και οικονομικά στις αραβικές χώρες στην Νότιο Μεσόγειο. Ένα πρόγραμμα που υπέγραψε ο Επίτροπος Φίλε, το μεγαλύτερο που υπογράψαμε ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νομίζουμε ότι είναι πολύ επίκαιρο, πολύ σημαντικό. Η περιφέρεια αυτή είναι μία από τις περιοχές προτεραιότητας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μας τις γυναίκες και χαρήκαμε διότι υπάρχει στενή εταιρική σχέση και θέλουμε να δώσουμε ορατότητα μεγάλη σε αυτό το πρόγραμμα, να το αναδείξουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα σημάνει αλλαγή για τις ζωές των γυναικών εκεί. Δουλεύουμε επίσης και πάνω σε άλλα προγράμματα τώρα ένα για την Ιγυρία, τη Βόρεια Ιγυρία, επίσης ε, σε ένα πρόγραμμα στη Γεωργία, άλλο στην Αίγυπτο. Ο προγραμματισμός μας διευρύνεται. Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο, εδώ αναφύονται διάφορα θέματα και ενισχύθηκε η συνεργασία μας. Σήμερα Μιλάμε για την προετοιμασία για την ε, Επιτροπή για την Κατάσταση των Γυναικών, αυτό. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας ε, για πολλές εκθέσεις και με άλλες επιτροπές όπου ε, συνεισφέρουμε και εμείς ή συνεισφέρουμε για παράδειγμα στη νέα ανακοίνωση για την κοινωνική προστασία για το Κοινοβούλιο, επίσης στις γυναίκες για τα Βαλκάνια, γυναίκες στην πολιτική λήψη αποφάσεων, οι γυναίκες στην κλιματική αλλαγή. Ε, υποβάλλουμε εκθέσεις και χαιρόμαστε για την ευκαιρία αυτή. Συνεργαζόμαστε επίσης με την κοινωνία των πολιτών εδώ στις Βρυξέλλες, διότι υπάρχει μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών που αφορά και τα θέματα ισότητας των φύλων και σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και όπως σας είπα, ε, όπου χρειάζεται συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη. Ε, με την Κυπριακή ή την Ιρλανδική Προεδρία για να συζητήσουμε για το δικό τους πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων. Αυτά είσαι ό,τι αφορά το έργο του γραφείου μας εδώ στις Βρυξέλλες. Πάω στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τι θα κάνουμε στις 25 Νοεμβρίου. Και αν έχετε ερωτήσεις για το έργο μας εδώ, ευχαρίστως να απαντήσω. Όπως κάθε χρόνο, οι UN Women οργανώνουν και συμμετέχουν σε σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τη Διεθνή ημέρα κατάργησης της βίας κατά των γυναικών. Φέτος, οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στο συγκεκριμένο πλαίσιο προετοιμασίας της 57ης Επιτροπής το Μάρτιο του 2013 για την κατάσταση των γυναικών με, ομάδα με θέματα προτεραιότητας την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών. Ως μέρος της εσωτερικής μας διαδικασίας προγραμματισμού θα κάνουμε ένα οδικό χάρτη για, με την εκδήλωση για την 27η Επιτροπή με πολλές δραστηριότητες για να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη, η κοινωνία των πολιτών, οι εμπλεκόμενοι, ούτως ώστε να υπάρξει συνένεση υπέρ της πολύ σημαντικής αυτής εκδήλωσης ε, της Επιτροπής για το Στάτους των Γυναικών της CSW. Τώρα, τι αποτέλεσμα θέλουμε να έχουμε στις 25 ε, Νοεμβρίου που θα γίνουν οι ορταστικέ εκδηλώσει, θέλουμε να καταδικάσουμε, να ε, γίνει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η βία κατά των γυναικών και κορισιών. Θέλουμε επίσης ε, να υπάρξει το, από τα κράτη-μέλη η άσκηση τη δέουσα επιμέλεια ούτω ώστε να ισχύουν όλες, όλοι οι κανόνε και θα πρέπει να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίε παντού για την πρόληψη και την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. Όπως ξέρετε, οι δύο τομείς προτεραιότητας για την CSW το Μάρτιο είναι η πρόληψη και τι υπηρεσίες προστασίας υπάρχουν ήδη και πώς μπορούν αυτές να γίνουν πιο συνεκτικές. Σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίες, εμείς θέλουμε στις 25 Νοεμβρίου να αρχίσουμε ένα νέο πρόγραμμα που λέγεται COMIT. Η κυρία Μπασελή θα κάνει μια θα απευθύνει πρόσκληση στα κράτη-μέλη και τους αρμόδιους υπουργούς για να αναλάβουν δέσμευση δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, να προστατεύονται οι γυναίκες ε, από τη βία κατά των γυναικών και να παρέχονται επίσης και υπηρεσίες. Ποιες θα είναι αυτές, ε, τι θα πρέπει να γίνει, να εγκριθεί καινούρια νομοθεσία, να υποστηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, να υπάρξει μια, ε, ένα κόκκινο τηλέφωνο για ενημέρωση. Υπάρχουν 16 ε, δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις που θα πρέπει να κοινοποιηθούν online, ούτω ώστε να δοθούν ενάβσματα σε άλλες κυβερνήσεις να κάνουν κάτι παρόμοιο. Και βέβαια εδώ χρειάζεται υποστήριξη από εσάς που είστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η υποστήριξή σας ε, ε, γιατί μπορεί να διαμεσολαβήσετε στις κυβερνήσεις σας να στηρίξουν το πρόγραμμα. Επίσης, θα, η κυρία Μπασιλή θα, ε, την ίδια μέρα θα κάνει μια δήλωση και ε, δήλωση βίντεο που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης θα γίνουν εκδηλώσεις σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο. Επίσης θα εορτάσουμε επίσημα στις 27 Νοεμβρίου το γεγονός αυτό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα ε, για την Ένωση για την Κατάργηση της Βίας. Ε, αυτή είναι μία και ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετέχει, η κυρία Μπασελή βέβαια, αλλά και η Μάρτζιν Καμάρα που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής για το Στάτους των Γυναικών φέτος για το 2013. Επίσης ε, υπάρχει το Celebrity και το Survival of Violence Against Women. Επίσης ε, θα ε, έχουμε την πορτοκαλή ημέρα όπου οι διάφορα δίκτυα νέων ε, και γυναικών θα προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν όλους τους παράγοντες σε εθνικό επίπεδο, να υπάρχει διαμεσολάβηση στις κυβερνήσεις για να ασχοληθούν και επίσης και οι ίδιοι θα οργανώσουν δραστηριότητες κατά της βίας ε, στις γυναίκες. Κάνουμε και περιφερειακές δραστηριότητες. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Αν θέλετε περαιτέρω ενημέρωση, ευχαρίστως να σας τη δώσω αργότερα. Όπως είπα όμως, η συνολική αιγίδα είναι η προετοιμασία για το CSW, οπότε το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε κατά το CSW να ανακοινωθεί κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις ε, για την 25η Νοεμβρίου. Ε, σε ό,τι αφορά το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η προετοιμασία για τη CSW. Η επιτυχία της CSW του χρόνου είναι κορυφαία προτεραιότητα για το UN Women. Οι UN Women έχουν ειδική εντολή να παρέχουν υπηρεσίες στην CSW. Το έργο μας πηγαίνει πέρα από τη γραμματιακή δουλειά. Ε, συνεχώς και ενάως δουλεύουμε για αυτά τα ε, θέματα σε διάφορα φόρα, ούτως ώστε να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση των γυναικών. Ε, του χρόνου η CSW θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν σε συμπεράσματα στη φετινή CSW και αυτό σοκάρισε πολλούς από μας, ιδιαίτερα διότι δεν ήταν ε, αμφισβητούμενο το θέμα της ενίσχυσης των γυναικών. Το επόμενο θέμα του χρόνου δηλαδή είναι η κατάργηση της βίας κατά των γυναικών και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, στην ατζέντα ενίσχυσης των γυναικών. Ε, ακόμα υπόκεινται σε οικογενειακή βία, στην οικογένεια, στο σπίτι, στις κοκκινότητες Πολύ συχνά υπάρχει σιωπή και ατιμορρησία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο σοβαρή έκφραση διακρίσεων και αποδυνάμωσης γυναικών και κοριτσιών. Άρα λοιπόν τι κάνουμε και πώς προετοιμαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως είπα, είμαστε η γραμματεία και παρέχουμε υπηρεσίες στο Προεδρείο, το οποίο είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για την ουσία ε, των εργασιών της CSW. Πρόσφατα κάναμε μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο Μπαγκόκ μαζί με έναν αριθμό οργανισμών του ΟΗΕ για να συμβάλλουμε και εμείς στις δύο εκθέσεις που θα ετοιμάσει η Γενική Γραμματέα για να ε, συζητηθεί από την CVSW. Όπως έμαθα σήμερα, η έκθεση έχει ανέβει τώρα ε, στην ιστοσελίδα, μπορείτε να τη δείτε online. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, διότι ε, δίνει τα πιο πρώτα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα συμπεριληφθούν αργότερα στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Δεύτερον, αρχίσαμε online συζητήσεις με 1.500 εμπλεκόμενους. Από τον Αύγουστο άρχισε αυτό, για να έχουμε απόψεις διαφορετικών απαντώντων ε, στις βασικές προκλήσεις και σε τρόπους αποφυγής της βίας. Η έκθεση επίσης είναι διαθέσιμη online, και μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα της CSW. E θα υπάρξει αυτή τη βδομάδα στο Λονδίνο μια συνάντηση οργανωμένη από την BFIT για να προετοιμάσει επίσης για τη CSW ο, η, κυρία Λάξμη Πούρη που είναι αναπληρώτρια γενική εκτελεστική διευθύντρια θα είναι παρούσα και θα κάνει μια δήλωση. Οργανώνουμε επίσης ένα φόρουμ των εμπλεκομένων μέσα Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο σκοπός αυτού του φόρουμ των εμπλεκομένων δεν είναι τόσο πολύ να εξετάσει τα θέματα ουσίας που θα συζητηθούν στη φετινή CSW, αλλά να σφυριλατήσει η πολιτική συνένεση που είναι η μείζον πρόκληση τώρα. Να φτάσουμε σε μια πολιτική συνένεση και να προχωρήσουμε έτσι και να καταλήξουμε στην φετινή συνάντηση CSW το Μάρτιο, να έχουμε συνένεση. Υπάρχει και μια συνάντηση ε, των γαλλόφωνων κρατών που οργανώνεται το Δεκέμβριο στο Παρίσι ε, και θα γίνει πρόσκληση και σε αφρικανικές χώρες πάλι για το σκοπό της συνένεσης. Οι UN Women μετέχουν στις σχετικές προετοιμασίες και ε, ήδη ε, πιστεύω, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό της γαλλοφωνίας και θα είναι πολύ σημαντικό θέμα για την CSW. Τώρα για τις δύο εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, η UN Women ε, καταρτίζει τις εκθέσεις. Η μία αφορά την πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών αντλώντας πάνω στις ορθές πρακτικές των κρατών μελών και τις τα αποτελέσματα των συναντήσεων των εμπειρογνωμών. Και το άλλο, η, άλλη έκθεση, αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Έχουμε μία για την πρόληψη, η άλλη είναι για την παροχή υπηρεσιών. Έτσι ορίζονται. Θα είναι έτοιμες πριν από το τέλος του χρόνου και μετά θα περάσουν από τη διαδικασία της μετάφρασης και θα είναι έτοιμη για την φετινή CSW. Επίσης, ε, Κάναμε πολύ, είχαμε πολύ στενή συνεργασία με τις, ε, τους διάφορους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, της οργανώσεις UNFPA, ε, UNICEF, παίζουν ρόλος για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε στη CSW. Ένα παράδειγμα τώρα τι κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο κάνουμε μια προσωμείωση, αν θέλετε, της CSW, ούτως ώστε να προετοιμάσουμε τους αντιπροσώπους, από την Ασία, από τις διάφορες χώρες, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για επιτυχής διαπραγματεύσεις ε, τον Μάρτιο. Εδώ στις Βρυξέλλες, λοιπόν, προσκληθήκαμε από, από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την DG Justice και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Γενική Διεύθυνση Ιδιοσύνης και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για να μοιραστούμε πληροφορίες και από κοινού να προετοιμαστούμε και είμαστε και πολύ ευγνώμονες στο Κοινοβούλιο για την ε, σημερινή πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό όλοι να συνεργαστούν για την επιτυχία της CSW. Ε, χαιρόμεθα διότι θα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή, όπως ελπίζουμε, θέση για την CSW και θα υπάρχει ενιαία προσπάθεια και προσβλέπουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου επίσης πάρα πολύ. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ως συμβολή για την CSW ε, ε, την ετήσια. Επίσης, ε, η Κυπριακή και η Ιρλανδική Προεδρία συμμετέχουν. Εμείς συζητούμε και θα συνεχίσουμε τον, και τον τους επόμενους μήνες να συζητούμε. Τώρα, κάποια θέματα ουσίας. Κοιτάω και λίγο. Μου δίνετε λίγο χρόνο ακόμα. Μου δίνετε. Ευχαριστώ. Καταρχήν είναι διαφυσβήτητο ότι τα φετινά αποτελέσματα από την CSW θα επιβεβαιώσουν πρότυπα και κανόνες για την κατάρριξη της βίας κατά των γυναικών. Υπάρχουν πολλοί κανόνες εδώ και πρέπει να τους αξιοποιήσουμε όλους. Είναι επίσης όμως σημαντικό το αποτέλεσμα να έχει μια διασύνδεση με πολιτικά πρότυπα και νόρμες σε άλλους τομείς. Πρέπει να γίνει μνήα στην πολιτική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών πρόσβαση στην παιδεία και στις οικονομικές ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Διότι η βία δεν συμβαίνει εν κενό, ενδογενώς συνδέεται με διάφορες μορφές διακρίσεων των, των φύλων σε, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική σφαίρα. Αυτή η διασύνδεση πρέπει να γίνει και θα πρέπει να υπάρξει ολιστική, ε, συνεκτική πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Δεύτερον, τα συμπεράσματα της CSW θα πρέπει να ζητήσουν επιταχυνόμενη και αποτελεσματική πρόληψη και αντίδραση. Είδαμε τα τελευταία χρόνια κάποιες πρόοδους. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν σειρά δράσεων, ε, ψήφισαν καινούργιες νομοθεσίες δέχτηκαν προγράμματα δράσης, τα ενέκριναν για να απαντήσουν και να αντιδράσουν στη βία. Τα προγράμματα και τα σχέδια δράσης πρέπει να χρηματοδοτούνται, να ελληνοποιούνται καλύτερα, να ε, παρακολουθούνται καλύτερα. Θα πρέπει να ε, υπάρξει πολυτομεακή ε, ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στα θύματα θα πρέπει να υπάρχει μια ε, νοοτροπία η οποία θα ε, καταδικάζει τη βία. Εμείς ε, έχουμε διάσπαρτες προσεγγίσεις, αλλά όχι συστηματικές, ολιστικές. Σε κάθε χώρα βλέπετε ότι γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το θέμα, αλλά χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης ότι υπάρχουν σαφείς διασυνδέσεις μεταξύ της πρόληψης, της βίας κατά των γυναικών και των αντιδράσεων και της προστασίας των θυμάτων. Και εδώ βέβαια είναι πολύ σημαντική ποινική νομοθεσία για τα θύματα αυτών των αξιόπινων πράξεων. Υπάρχουν πολλές, πολλά υποσχόμενες πρακτικές και σε αναπτυσσόμενες χώρες που ξεπερνούν την ευαισθητοποίηση ε, και συμπεριλαμβάνουν την συμμετοχή ανδρών και ε, αγοριών, πολύ σημαντικό, και τους θρησκευτικού ηγέτες. Εμείς δουλεύουμε πολύ ως UN Women με τους θρησκευτικού ηγέτες χωρών, ελπίζοντας σε μια αλλαγή. Η επόμενη συνεδρία της CSW e θα είναι καλή ευκαιρία για να συλλέξουμε αυτές τις καλές πρακτικές, να έχουμε προληπτικές στρατηγικές που θα αυξήσουν την προστασία των γυναικών, για να σταματήσει η βία στις ρίζες της και να υπάρξει και συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων. Ε, Επίση, θα πρέπει τα αποτελέσματα να αναγνωρίζουν φέτο ότι υπάρχουν πολλέ μορφέ βία. Ε, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, ε, γάμοι παιδιών ε, και πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλές μορφές, πρέπει όμως να αναγνωριστεί ότι η πιο διαστραμμένη μορφή βία είναι η οικογενειακή ε, από μέλη της οικογένειας ε, όπου γίνεται σε πολλές ε, περιοχές του κόσμου και οδηγεί σε τραυματισμό ψυχολογικό και πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Τέλος, τα συμπεράσματα πρέπει να τονίζουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και θέμα που αφορά την ανάπτυξη, ε, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη. Ε, αποτελεί μεγάλο βάρος στις, κοινωνικές, οικονο... Ε, εθνικές οικονομίες. Ε, υπολογίζεται σε 33 δις δολάρια είπα. Για όλα αυτά η καπάλυψη της βίας θα πρέπει να είναι κομμάτι κάθε δείκτη για την, ε, ε, τα δικαιώματα και την ισότητα των γυναικών και θα πρέπει να είναι και ε, συμπεριλαμβάνεται στο αναπτυξιακό πλαίσιο του 2015. Δύο λόγια ακόμη για τις στρατηγικές διαπραγματεύσεων. Πώς θα προετοιμαστούμε για την επιτυχία, ανέφερα ορισμένα πράγματα, συνεχιζόμενες δραστηριότητες κλπ αλλά είναι αναντήρητο ότι η προώθηση της ισότητας των γυναικών και η ενίσχυση των γυναικών αντιμετωπίζει ε, κάποια προβλήματα. Ε, το περιβάλλον παλαιότερα ήταν λίγο πιο αισιόδοξο, ε, ήταν πιο οραματικό. Τώρα πολλοί παράγοντες και συνθήκες ασκούν πιέσεις στην πρόοδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Τονίζω ότι δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή τα προβλήματα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι οικονομικές, δημοσιονομικές πιέσεις επηρέασαν την κατάσταση των γυναικών στις αναπτυσμένες χώρες. Η πολιτική κρίση, οι οικονομικές, κοινωνικές στάσεις και εξελίξεις επίσης έπαιξαν τον ρόλο τους. Ε, αυτό, αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε με προσοχή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε μεταξύ των ε, αναπτυσσόμενων ε, πρωτοπόρους που θα τους αξιοποιήσουμε. Ε, πολλές από τις χώρες σας έχουν διμερείς σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι σχέσεις αυτές. Υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας και υποστηρίζουμε, όπως είπα και πριν, σε μια ενιαία ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση είναι να έχουμε μια ισχυρή ε, ουσιαστική βάση, αντικειμενική. Αυτό το κάνουμε με υψηλή ποιότητα εκθέσει για θέματα προτεραιότητα από, τη Γενική Γραμματεία, ε, από τη Γραμματεία και προπαρέχοντα τεχνικέ υπηρεσίε πριν και κατά τη διάρκεια των συνόδων, των συνεδριάσεων. Επίση, ε, θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στα λεπτά θέματα, όπω δικαιώματα των γυναικών στην αναπαραγωγική σεξουαλική υγεία ε, τα δικαιώματα στον τομέα αυτά, αυτών αποτέλεσαν επίμαχο θέμα μεταξύ των αντιπροσωπιών. Ε, υπάρχουν διαφορές ε, στις πρακτικές, αλλά η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα είναι σημαντικά για την ενίσχυση των γυναικών. Και αυτό αναγνωρίζεται από πολλά έγγραφα. Ε, θα πρέπει να διαλύσουμε το μύθο γύρω από τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα και τι σημαίνουν όλα αυτά. Ε, ισχύει αυτό κυρίως για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε τα πρότυπα που υπάρχουν και δουλεύουμε πολύ στενά με την ε, UNFPA για αυτά τα θέματα σε ό,τι αφορά ε, τι μπορούν να κάνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να στηρίξουν τις διαδικασίες αυτές. Όπως προανέφερα, χαιρετίζουμε και προσβλέπουμε σε συνεργασία με, τις, με σας και τις, μέσω ημών με τις εκλογικές σας περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί για να στηρίξουμε μια ε, στιβαρή θέση της Ένωσης, να στηρίξουμε, ε, αναφέρατε και τη Ρωσίδα Μανσού που ζήτησε αυτή την ε, παγκόσμια νέα σύμβαση, το χαιρετίζουμε αυτό, ήταν σε ένα πάνελ με την αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια πέρσι, την περασμένη εβδομάδα που ετέθη το θέμα και η UN Women συμφώνησε με τις προτάσεις αυτές. Ε, μακάρι να είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα από την CSW. Και όπως είπα, το νέο πρόγραμμα Commit που έχουμε, καλό θα ήταν να υποστηριχθεί από εσά. Γιατί η Διεθνή Μέρα για τα Κορίτσια. Μπορούμε να το πούμε αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εντάξει, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Όχι, θα μιλήσω σε ειδικά. Δεν θα αλλάξω για τα αγγλικά. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσίαση στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και πραγματικά είσαστε, ε, η υπηρεσία σας είναι σημαντικός εταίρος της Επιτροπής Γυναικών του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στους δύο θεσμούς και σίγουρα και στη μελλοντική μας συνεργασία θα φανεί αυτό ακόμη σαφέστερα. Θα ήθελα τώρα να αρχίσει η συζήτηση. Ε, η κυρία Μορβάη θα πάρει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Η βία κατά των γυναικών έχει ενταχθεί στην στο θεματολόγιο των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω από το 1990. Ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια. Αναφερθήκατε σε εμπόδια που υπάρχουν παντού. Είπατε ότι δεν είναι γεωγραφικά τα εμπόδια αυτά. Θα νόμιζε κανείς ότι όλοι συμφωνούν, ανεξαρτήτως πολιτικών προτεραιοτήτων, ότι ο βιασμός, η παρενόχληση των γυναικών είναι κάτι λάθος είναι λάθος. Γιατί λοιπόν οι κυβερνήσεις, τα νομικά συστήματα, σε συστήματα απονομής δικαιοσύνης, οι αστυνομίες δεν, δεν καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να απαλείψουν ένα φαινόμενο το οποίο όλοι συμφωνούν ότι είναι θεμελιακά λάθος. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα standards, ε, κάποια ελάχιστοι κανόνες ε, ε, κάποια ελάχιστα κατώτατα νομικά όρια, εχέγγυα, δικαιώματα κτλ. Δεν έχει έρθει ο χρόνος να αναπτύξουμε κάποιες ελάχιστες εγγύησεις και στον τομέα της βίας κατά των γυναικών. Τι είδους νομικά δικαιώματα θα έπρεπε να έχουν, για παράδειγμα, οι... εκείνες που επιβιώνουν από την οικιακή βία τι είδους υπηρεσιών δικαιούνται, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Τι άλλες υπηρεσίες οφείλουν οι κυβερνήσεις να παρέχουν στα θύματα της βίας, της οικιακής βίας. Ε, νομίζω ότι να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εγγύησεις ε, θα διευκολύνουν όλους τους φορείς που ενεργοποιούνται, τον ΟΗΕ και τα λοιπά, να αξιολογήσουν καλύτερα το καθεστώς, ε, το, το πού βρίσκεται η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών και η καταπάτηση των η προστασία από την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θα σε ευχαριστούμε. Ε, σύντομη παρέμβαση, σύντομες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να δώσετε το παράδειγμα, νομίζω. Να σας μιμηθούν κι άλλοι. Και τώρα η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Γυναικών και εγώ εκπροσωπώντας τους πράσινους θα ήθελα και εγώ να σας ε, καλωσορίσω. Αναφέρετε κάποια θέματα εκπαιδευτικά. Όπως είπατε πέρυσι ή μάλλον φέτος η CSW δεν κατάφερε να καταλήξει σε κοινό ανακοινοθέν. Ε, ε, μου φαίνεται φρικτό αυτό. Και μιλήσατε για την για το γιατί δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό και να βρεθούν άνθρωποι που να προάγουν τον αγώνα αυτόν στις ε, μη αναπτυσσόμενες χώρες εσείς πώς θεωρείτε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βρεθούν κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες ε, που να προάγουν το έργο της προετοιμασίας του συνεδρίου αυτού. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια κοινή θέση την οποία μπορεί να εκφράσει η πρεσβεία της, Ενω... της Ενωμένης Ευρώπης. Ε, γιατί βέβαια το κάθε κράτος μέλος κάνει τα δικά του. Αλλά εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκή στήριξη για αυτό που ζητάτε ή βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα και εκεί. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω. Η όλη διαδικασία υπάρχει εδώ και 10 χρόνια όπως είπατε. Ποιες ήταν, υπήρξε επιτυχής. Ε, καταρχήν έφερε κοντά όλους τους διαφορετικούς φορείς, ε, πράγμα που δεν είναι και εύκολο βέβαια. Επίσης, είχε κάποιον θετικό αντίκτυπο εντός του ευρωπαϊκού συστήματος. Το ελπίζω. Εκτός του ευρωπαϊκού συστήματος είχε κάποιο θετικό αντίκτυπο και ο κ. Μπατσελέ το, το είπε. Ποια ήταν τα ωφέλη. Ε, σήμερα θα ψηφίσουμε το θέμα της καταπολέμησης των στερεότυπων των φύλων. Μιλούμε για στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύω τα στερεότυπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, έχετε ασχοληθεί και με αυτό, γιατί νομίζω ότι χωρίς αυτό ε, φυσικά χρειαζόμαστε όλα τα άλλα, προστασία, νόμους λοιπά. Αλλά αν δεν αλλάξουν τα στερεότυπα, ε, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που προσλαμβάνεται η γυναίκα και η νεαρή κοπέλα, το κορίτσι, δεν θα γίνει τίποτα. Και τέλος, για τις ομοφιλόφιλες γυναίκες. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ επίμαχο ζήτημα, πολύ ακαθόδες ε, εργάζεστε καθόλου πάνω στα δικαιώματα των ε, λεσβιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κώστα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτήν την απόφαση ε, της αυτή την απόφαση να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς σχετικοί με τις γυναίκες εδώ στις Βρυξέλλες ε, θα υπήρξε και μια επίσκεψη στην την Ισία. Υπάρχει και ένας φορέας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια για τις γυναίκες. Είπατε ότι μία από τις προτεραιότητες της δράσης σας, του προγράμματός σας, αφορά ακριβώς τις γυναίκες της Νότιας Μεσογείου. Θα ήθελα να έχω την εκτίμησή σας. Εμείς έχουμε κάνει μια δουλειά στην Ισία. Ξέρουμε ότι και το Μαρόκο, έχει κάποιο γραφείο ε, και στην Λιβύη νομίζω δεν έχετε καταφέρει να ανοίξετε κάποιο γραφείο. Ε, και είναι ίσως και οι πληροφορίες που έχουμε λίγο συγκεχημένες. Εγώ προετοιμάζω μια έκθεση πάνω σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίες που να μας ε, δείχνουν λίγο πώς έχει η κατάσταση. Όσο αφορά την βία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον ε, Μάρτιο κάνει σημαντική δουλειά. Έχουμε προετοιμάσει ένα πακέτο ολόκληρο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ε, ξέρω ότι στις 25 Νοεμβρίου θέλει να ε, απευθύνει αυτή την έκκληση η κυρία Μπατσελιέ. Προσοχή όμως, γιατί ένα φαινόμενο που είναι ένα αδοικό φαινόμενο, τουλάχιστον στην δική μου χώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα καταδίωξης, αν θέλετε, ε, καταδίωξης γυναικών ε, από την πρώην οικογένειά τους. Έχουμε 100 τέτοια περιστατικά στην ε, Ιταλία. Έχει, ε, έχει αλλάξει λίγο το πρόβλημα ή μια όψη του προβλήματος. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς έχει η προστασία των, της συγκεκριμένης κατηγορίας γυναικών διεθνώς. Τώρα για τα θύματα της σεξουαλικής βίας. Ε, θα πρέπει στο θέμα αυτό να υπάρξει και μια πρόληψη ε, των δυσκολιών που συναντούν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια τούτο και του. Ε, και, και τα προβλήματα της βρεφικής θνησιμότητας, της νεογνικής θνησιμότητας. Φυσικά αυτό είναι κομμάτι του οικογενειακού προγραμματισμού, εντάξει, αλλά καμιά φορά χρειάζεται ε, και ένα άλλο είδος προγραμματισμού και αυτό μας το επισημαίνουν ιδιαίτερα οι γυναίκες της Νοτιού Μεσογείου ε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και της θνησιμότητας που αντιμετωπίζουν κατά τον τοκετό. Ευχαριστώ. Ε, don't have any more Δεν βλέπω να, υπάρχει, να υπάρχουν άλλοι ομιλητές προς το παρόν. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Vad σου vi bli eh, på? Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια μόνο. Όπως είπε και η κυρία Μορβάη, πρέπει να ασχοληθούμε με τα ελάχιστα πρότυπα. Στην Επιτροπή θα συζητηθεί αυτή η οδηγία για την θέσπιση ελαχίστων προτύπων και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Τώρα σας κάνω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Όταν εξετάζουμε το θέμα της ε, νέας σύμβασης ε, για τον ΟΗΕ. Σκεφτόμαστε και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, ε, που καλύπτει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες, ε, αλλά πιο συγκεκριμένα όπως είπε και η κυρία Λούνατσεκ υπάρχουν και ελλείψεις, αλλά ε, κατά τη διαστολή καλύπτονται σημαντικά ζητήματα και μια τέτοια διεθνή σύμβαση είναι το προσφορότερο εργαλείο για την ε, μονάδα του η απασχολείται με τις ε, γυναίκες. Ε, θα πρέπει λοιπόν, αν θέλετε, να μας σχολιάσετε και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θα μπορούσατε λοιπόν να πάρετε το λόγο, αν θέλετε, για να σχολιάσετε τις παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Σχετικά με το πρώτο θέμα, δηλαδή ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποια είναι, είναι τα βασικά προσκόμματα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τομείς ε, και θα αναφερθώ μόνο σε έναν. Ε, το θέμα του, του οικογενειακού βιασμού, συζυγικού βιασμού, ε, είναι ένα από τα προεξάρχοντα θέματα και στις ε, ε, φετινές συζητήσεις μας θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και υπάρχει ομολογουμένως διάσταση απόψεων για το ζήτημα αυτό. Για τα ελάχιστα πρότυπα, για να απαντήσω και στους δυο σας, ακριβώς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που δηλώνεται ότι είναι ένας από τους στόχους εδώ στην Επιτροπή των Γυναικών, διότι η πρωτοβουλία Αυτό αυτόν ακριβώς το στόχο έχει. Το πέρυσι ε, ξεκινήσαμε με τις 16 δράσεις που εισηγήθηκε η κυρία Μισελ Μπασελέ για να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα σε ένα πακέτο που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες, ελάχιστη πρόνοια και πρόληψη, σχετικές δράσεις και στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ε, ο στόχος είναι να έχουμε μια ολιστική, μια σφαιρική προσέγγιση για το ζήτημα που υπερβαίνει τις οποιασδήποτε εθνικές πρωτοβουλίες. Έτσι θα ε, διαμορφώσουμε ένα πακέτο βασικών υπηρεσιών προς τις γυναίκες θα γίνει ανταλλαγή απόψεων ε, για το θέμα των ελαχίστων πρότυπων, ανταλλάξουμε απόψει για τον ορισμό των ε, ελαχίστων πρότυπων Καταρχά. Ε, καλό θα ήταν να συνεργαστούμε στενότερα με την Επιτροπή σας για αυτό το θέμα. Ε, ως προς το ερώτημα της κυρίας Λούναντσεκ για τα στρατηγικά ζητήματα και πόσο ε, ποια ομοφωνία υπάρχει στη μονάδα του ΙΕ για αυτά τα ζητήματα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της CSW. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο αναπληρωτή διευθυντής μας ήρθε στις Βρυξέλλες ε, την περασμένη εβδομάδα. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα και συγκεκριμένα η προετοιμασία για την επόμενη σύσκεψη τη CSW. Έχουμε τον κύριο Λαμπρινίδη που είναι ο νέο ειδικό ε, εκπρόσωπος ε, συνεργαζόταν δικαιοσύνη με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκάθαρα προωθεί αυτά τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτές τις δράσεις. Παρόλα αυτά, που απέχουμε από την συνενετική λύση. Όμως υπάρχει μία ομοψυχία και όλοι τίνουν προς μία συνενετική θέση. Συζήτησα και με εκπροσώπους της Κυπριακής και της Ιρλανδικής Προεδρίας και διαπιστώνω ότι υπάρχει πολιτική βούλη σε σημαντικό βαθμό για να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή θέση. Δεν την έχω δει ακόμη και δεν ξέρω πόσο ισχυρή θα είναι, αλλά πάντως από τους Ιωνούς ε, ε, θα έλεγα ότι θα είναι μάλλον θετική έκβαση και είμαστε αισιόδοξοι. Ε, ως προς ε, το, ε, την επιτυχία της δράσης μας και το πώς επηρεάζουμε το σύστημα του ΟΗΕ. Κοιτάξτε, ο Γενικός Διευθυντής ε, κατά την σύσταση της Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι η θέσπιση αυτής της μονάδας δεν απεκδεί των ευθυνών του στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Η κυρία Μπασελή είπε ξεκάθαρα, εγώ δεν θέλω να είμαι μια αστυνομία για τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων από κοινού με το σύστημα και το σχέδιο δράση του ΟΗΕ καταλήξαμε σε πολύ συγκεκριμένε δράσει για την πρόθεση των ζητημάτων ισότητα των δύο φύλων στο εσωτερικό του συστήματο ε, του θεσμικού συστήματος του ΟΗΕ και αυτό το σχέδιο δράσης συζητήθηκε για κάποιου μήνες, εγκρίθηκε και τώρα ε, πιστεύω ότι συνιστά μια πολύ καλή πρακτική και όντω αναβαθμίζει την ε, ενδοϊπηρεσιακή συνεργασία στον ΟΗΕ για τα θέματα που ε, άπτονται των γυναικών. Οπότε ακολουθούμε μια θετική τροχιά και ε, τα αποτελέσματα, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και λειτουργούν καλύτερα συντονιστικοί μηχανισμοί. Όντω, ε, αυτό είναι και μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητε τη εντολή που έχει η μονάδα μα. Δεν υπήρχε καν αυτό προηγουμένω. Ε, προτού συσταθεί η μονάδα μας, ποτέ δεν είχαμε αρκετά υψηλό εκπρόσωπο που να επιλαμβάνεται αυτό τον ζήτημα τη ισότητα των δύο φίλων που μπορεί να μετάσχει στα τα πολιτικά φόρα του συστήματος του ΟΗΕ, διότι η κυρία Μπασελέ είναι παρά του Γενικού Γραμματέα ε, του ε, ΟΗΕ και ως εκ τούτου μετάσχει σε όλες τις συζητήσεις ε, που αποσκοπούν στο συντονισμό της ενδοπηρεσιακής δράσης του ΟΗΕ για τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων, οπότε εισακούεται η κυρία Μπασελέ. Ε, τώρα θα συμφωνήσω μαζί σας για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το θέμα ε, της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται στις γυναίκες ε, και στα κορίτσια ανά τον κόσμο. Έχουμε τα στερεότυπα, παραδείγματο χάρη για τη, τα δύο φύλλα, ότι δεν πρέπει να μετάσχουν στη Βουλή, να είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων οι γυναίκε, παραδείγματο χάρη. Ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα στερεότυπα σε διάφορε χώρε. Για το ζήτημα των λεσβιών, όντω είναι ύψιστη προτεραιότητα και ο Γενικό Γραμματέα αναφέρθηκε στα δικαιώματα ε, των ομοφιλοφίλων έκανε μια πάρα πολύ ισχυρή δήλωση για το ζήτημα, διότι έγινε πρώτον στο ανώτατο επίπεδο του ΟΗΕ, αλλά φετέρου εφόσον προέρχεται από τον Γενικό Γραμματέα, εισέρχεται παρισφρή αυτό το βήμα σε όλες τις ε, δομές ε, του ΟΗΕ για την ε, Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή υλοποιούμε την αναθεώρηση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής. Αυτός είναι ο τίτλος μιας άσκησης ε, που επιχειρούμε για να ενισχύσουμε τις ε, επιτόπιες δυνατότητες που έχουμε, τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για τον οργανισμό μας. Ε, αυτή είναι μείζον πρόκληση ορισμένες φορές για την ε, μονάδα μας, ε, διότι η χρηματοδότηση και τα κονδύλια δεν ε, είναι στο ύψος των απαιτήσεων και των προσδοκιών που έχουν όλοι από τη δράση της υπηρεσίας μας. Το εκτελεστικό μας συμβούλιο θα εξετάσει αυτό το ζήτημα ε, πριν το τέλος του έτους και θα διαπιστώσει που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητές μας ε, στην Νότιο Μεσόγειο και συγκεκριμένα ένα ενδεχόμενο είναι η σύσταση γραφείου στη Λιβύη. Στο Κάιρο εσχάτως έγιναν τα εγγένεια ενό περιφερειακού γραφείου και η νέα περιφερειακή διευθύντρια ήρθε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα με τη νέα αναπληρώτρια διευθύντρια της μονάδας μας ε, και όντως ε, και αυτά συνιστούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά θέσατε και το ζήτημα της θέσπισης διεθνών προτύπων. Αναφέρθηκα ακροφυγώς αυτό, δηλαδή το πώς θα ε, χειριστούν τα κράτη-μέλη αυτό το ζήτημα μεμονωμένα. μονόμενα θα απαντήσω και πάλι ότι όντως πρέπει να θεσπιστούν κάποια ελάχιστα πρότυπα και κατανοώ το ερώτημά σας για τα διάφορα είδη βίας, την παρακολούθηση, παρενόχληση κτλ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη βίας, όχι να επικεντρωνόμαστε σε ένα, ναι, να ασχοληθούμε με την επίμονη και επώδυνη παρακολούθηση, την παρενόχληση και ούτω καθεξής. Um, Για το θέμα της αναπαραγωγικής υγείας, ε, το θέμα της πρόληψης ε, είναι πηγή μεγάλων ανησυχιών. τώρα για την τροπο... αλλαγή των νοοτροπιών των γυναικών και των κοριτσιών, ε, κυρίως η UNF USPA και η UNICEF ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα κυρίω, αλλά το θέμα τη πολιτική για την κατάρτιση πολιτική και η προώθηση των συμφερόντων μα το υπονομαζόμενο advocacy, είναι ζητήματα που απασχολούν την μονάδα μα. Μιχαήλ, ε, με ρώτησε και εσύ για τα ελάχιστα πρότυπα, το σε αυτό και χαιρόμαστε για τη μελλοντική συνεργασία μα για αυτό το ζήτημα. Α, για αυτή τη νέα σύμβαση που ρώτησε. Ε, Όντω ε, θα εξετάσουμε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ε, ελπίζουμε ότι σύντομα θα ακυρωθεί. Υπάρχουν όμως και άλλες συμβάσεις στη Λατινική Αμερική, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν καλά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές που, από τα οποία μπορούμε να εμπνευστούμε. για να διαπιστώσουμε ποιο είναι ο προσφορότερο τρόπος για να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Πρόκειται για μια νέα πρόταση και όλα θα είναι συνάρτηση των συζητήσεων και των εξελίξεων. Πάντως, οποιαδήποτε υποστήριξη από πλευρά σα είναι ευπρόσδεκτη και σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Κυρία Λούνατσεκ. Thank you uh, Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο, γιατί κάτι θυμήθηκα που το ξέχασα την πρώτη φορά που ζήτησα το λόγο. Πρόσφατα υπήρξε ένα πρόβλημα με τις οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με την πρόσβαση των συζητήσεων στη διάσκεψη CSW ε, και αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των μελών των μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορούν να συμμετέχουν. Ε, πώς το βλέπετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό στον τομέα αυτό όπως και σε άλλους τομείς να έχουμε διαπιστευμένα άτομα τα οποία να μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις με τις κυβερνήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής που ενδεχομένως θα ήθελε να παρέμβει με μια σύντομη ερώτηση. Θέλει κάποιο να πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μήπω, Θέλει κάποιο ε, οποιοδήποτε να πάρει το λόγο. Όχι καλά. Σα ξαναδίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ Τσέκ για αυτή την τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους στη Νέα Υόρκη υπάρχει στενή συνεργασία με το Bureau για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην κοινωνία των πολιτών. Η κυρία Μπατσελιέ ε, συναντήθηκε για πρώτη φορά με μια συμβουλευτική επιτροπή των ΜΚΟ, ε, την οποία συνέστησε. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν από δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη. Υπήρχαν εκεί εκπρόσωποι από ΜΚΟ από όλο τον κόσμο, από το λόμπι των γυναικών. Υπήρχαν και άτομα εδώ από τη σκηνή των Βρυξελών. Συζητήθηκε το θέμα και εκεί και θα κάνουν ό,τι μπορούν ε, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών ε, θα έχει ικανή πρόσβαση. Γιατί να έχουμε ισχυρή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών και είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της CSW ότι δεν υπάρχουν μόνο κράτη παρόντα, αλλά ότι μετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Πραγματικά το σημειώνω και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να διευκρινίσω το θέμα αυτό ενώπιον των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ε, ίσως ε, Είχα υποσχεθεί να πω λίγα λόγια και για τον ε, διεθνές καθεστώς των νεαρών κοριτσιών. Δεν το έχω κάνει. Φέτος στις 11 Οκτωβρίου έγινε η ε, ε, ε, για πρώτη φορά γιορτάσαμε το Διεθνές Έτος Νεαρών Κοριτσιών εδώ στις Βρυξέλλες. Συνεργαζόμαστε με το Plan International και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και οργανώσαμε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, ασφαλώς θα το ξέρετε. Σε παγκόσμιο επίπεδο εργαζόμαστε με την UNICEF, την UNFPA, και υπάρχει και ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για, τη, για τους γάμους μεταξύ παιδιών. Ε, στο πλαίσιο αυτού του πάνελ έτσι δώσαμε περισσότερη προσοχή στα νεαρά κορίτσια, στο θέμα του γάμου μεταξύ παιδιών και της προσπάθειάς μας να απολύψουμε αυτό το φαινόμενο. Χαίρομαι που το θέμα αυτό συζητείται όλο και περισσότερο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το εκτιμούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που πραγματικά χρήζει περισσότερη ε, προσοχής και αν υπάρξει κάποιο ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν πολύ καλό. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ανταλλαγή απόψεων αυτό το πρωί. Αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις παρακαλώ ε, ελάτε να μας δείτε στο γραφείο μας εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε και πάλι. Όπω σα είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, χαιρόμαστε όλου ιδιαίτερω που ήρθατε στο Κοινοβούλιο και επιθυμούμε να συνεχιστεί αυτή η τόσο καλή συνεργασία με τη μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες, γιατί πρόκειται για δύο παρεμφερή ε, ε, θεσμικά όργανα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικεντρώνετε την προσοχή σας ακριβώς σε αυτό το θέμα της βίας ε, κατά των γυναικών ε, και τονίζουμε πόσο επιτακτικές είναι οι ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα λόγω της ε, χαρακτηριστικής έλλειψης μέτρων. Χαιρόμαστε λοιπόν διότι συνιστά προτεραιότητα και για μας αυτό το θέμα το θέμα της βίας και το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσδώσουμε μια ισχυρότερη πολιτική διάσταση ε, σε αυτό το θέμα της βίας των αντρών κατά των γυναικών. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία που δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο ε, φαινόμενο. Πλήττει τις γυναίκες σε όλους τους τομείς και καθημερινό. Και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τη, αυτά τα ζητήματα μέσα από δομές που υπάρχουν όπως η Επιτροπή μα και η μονάδα σα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συνεργασία μας από πολλές πλευρές και ε, εν ώψη της συνεδρίασης του CSW καλό θα ήταν να ξανασυζητήσουμε για να δούμε ποιες συγκεκριμένες δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε. Ε, θα ε, σας ε, προσκαλέσουμε και πάλι στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας ημέρα. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, δηλαδή σημείο 6, ενημέρωση από το ταξίδι της Επιτροπής μας, την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που επισκέφθηκε την, την Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κώστα που είναι η συγγήτρια για την έκθεση που θα καταρτήσουμε. μάλλον το σημείωμα που θα συντάξουμε για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, η Τινησία είναι μια χώρα όπου, που έχει καλό σκορ, θα το έλεγα έτσι, στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. 27% των βουλευτών είναι γυναίκες. Μην ξεχνάτε τι γινόταν στον καιρό της δικτατορίας πολλά ε, ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν 27% των ε, βουλευτών γυναίκες. Επίσης, πολλές δράσεις που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναίκων, ανισότητες στους μισθούς, προστασία των δικαιωμάτων αναπαραγωγικής υγείας, καταπολέμηση της βίας έχουν αναλυφθεί από την Τινησία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Πήγαμε εκεί σε μια συναρπαστική περίοδο μετά την Αραβική Άνοιξη. Ε, και ε, το μείζον, ε, το φλέγον θέμα είναι το θέμα του συντάγματος και γι' αυτό δυσκολευτήκαμε να σχολιάσουμε όλα τα ζητήματα διότι όλα ασχολούνται με αυτό ακριβώς το ζήτημα για κάποια συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος σχετικά με την οργάνωση του πολιτικού βίου και ότι αν ε, δεν ε, ευοδοθούν οι προσπάθειές τους, μας είπαν για κάποια από αυτά τα άρθρα, τότε θα πληγούν τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Ε, διαπίστωσα ταυτόχρονα ότι σε επίπεδο Βουλής γίνεται πολύ ανοιχτή συζήτηση. Δηλαδή όλα τα πολιτικά κόμματα μέσα στη Βουλή συνεργάζονται ε, και συζητούν άνοιχτα για αυτά τα ζητήματα. Ορισμένες φορές ε, χρειάζεται κανείς να οπισθοχωρήσει για να κάνει ένα άλμα ε, στη συνέχεια. Θα δούμε ποιες, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται ανοιχτή συζήτηση. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Λοιπόν, μετά από αυτά τα σύντομα εισαγωγικά σχόλια, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα, που είναι και η συγκήτριά μας για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία και οι συναντήσεις που είχαμε υπήρξαν πολύ σημαντικές. Ιδίω για να ενημερώσω τους συναδέλφους, ιδίω με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Ενώσης των Γυναικών, και μεταξύ όλου του φάσματος των απόψεων, αλλά και με τους συνομιλητές μας, τους πολιτικούς, UN ε, ε, Γυναίκες, Παγκόσμια Τράπεζα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για την μικροπίστοση που μας έδωσε και ιδέες. Ε, είναι σαφές ότι στο πλαίσιο της έκθεσής μου όχι μόνο για την κατάσταση των γυναικών και στις τέσσερις χώρες που θα περιλάβουμε. Στις τέσσερις αυτές χώρες η Τινησία έχει μια εμβληματική θέση. Είναι μια χώρα η οποία έχει μια ιστορία και ένα καθεστώς που σε 40 χρόνια. Παρόλα αυτά όμως σε σχέση με άλλες Ισλαμικές χώρες ε, η κατάσταση, ο προσωπικός κώδικας, ε, τα δικαιώματα των γυναικών είναι αρκετά προηγμένα σε σχέση με άλλες χώρες όπως είπα. Υπάρχει ήδη μια παρουσία στο Κοινοβούλιο σημαντική, στο άνω και στο κάτω νομοθετικό σώμα. Υπάρχει μια μεγάλη ζωντάνια της κοινωνίας των ε, πολιτών, το γυναικείο κομμάτι της, πολλές γυναίκες επιχειρηματίες, πολλές ε, καθηγήτριες πανεπιστημίου, ε, μια σημαντική παρουσία των γυναικών. Φυσικά είδαμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά και από όλες τις μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε ότι υπάρχει μια διαφορά έντονη από κοινωνικο-οικονομική άποψη ε, και από άποψη ουσιαστικής ισότητας. Επίσης μεγάλη διαφορά μεταξύ του Βορρά και του Νότου, μεταξύ των πόλεων και της Υπέθρου. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άλλοι ε, συνάδελφοι, αλλά εγώ προσωπικά είχα λόγους να ελπίζω και λόγους ε, να ανησυχώ σοβαρά. Ε, νομίζω ότι συμβαίνουν εκεί μεγάλες αλλαγές. Η συγκέντρωση της προσοχής των γυναικών έχει, βρίσκεται βρίσκεται εν εξελίξη κατά κάποιον τρόπο. Θυμάστε τις μεγάλες διαδηλώσεις για το άρθρο περί της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και της συμπληρωματικότητας του γυναικού και του ανδρικού ρόλου. Ε, αυτό έχει δείξει ότι υπάρχει μια πίεση της διεθνούς και της εθνικής κοινή γνώμης και πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν και να προάγουν το ζήτημα περισσότερο. Τώρα όσο αφορά για, τα διάφο για τις διάφορες πολιτικές πλευρές, ε, θεωρώ σημαντική τη συμμαχία που υπάρχει με πολλούς δημοσιογράφους ε, και με τις επαγγελματικές οργανώσεις ε, των δημοσιογράφων που έχουν έτσι στη διάθεσή τους σημαντικά μέσα ε, και είναι καλό η Ευρώπη, οι βουλευτές, να μην τους αφήσουμε μόνους του, μόνες τους σε αυτή τη διαδικασία, να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις. Αυτός είναι λόγος για να ελπίζω βέβαια, δεύτερος λόγος για να ελπίζω. Υπάρχει, πώς να το θέσω, νομίζω ότι η πλειοψηφία των γυναικών που συναντήσαμε Ε, οι Τινήσιες δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο παρελθόν. Ε, η συνάντηση με τους βουλευτές ε, είναι 60 οι γυναίκες το... στο νομοθετικό σώμα εκεί. Ή την Ισία ή η την η, η η συμμαχια των Κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία. Ε, υπάρχουν δύο κόμματα. Ένα είναι καθολικοί σοσιαλδημοκράτες, ε, ε, ρεπουμπλικάνοι, πιο λαϊκό κόμμα. Η αίσθηση λοιπόν είναι, όπως το έλεγε και ο πρόεδρος, ότι υπάρχει μεγάλη επίγνωση μεταξύ των γυναικών ε, για το θέμα ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των μετριοπαθών Ισλαμιστών και των άλλων δυνάμεων της κοινωνίας, διαφόρων πολιτικών χριών, να βρεθεί λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ μιας τινήσιας ταυτότητας και των θεμάτων της καθολικότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ε, ε, κατοχήρωσης ε, των γυναικείων δικαιωμάτων στο Σύνταγμα, το θέμα της ισότητας, μια επιθυμία να διατηρηθούν τα αποτελέσματα που επετεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια προς το καθεστώς των γυναικών. Μέσα στο Σύνταγμα θέλουν να υπάρξει σαφής επίκληση της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι ώστε να περάσουν και στο εσωτερικό δίκαιο. Υπήρξε και ε, ε, ενώ το άρθρο 1 του συντάγματος προβλέπει μία αποδεκτή προσθήκη καρπός μεγάλων προσπαθειών το κράτος της Τουνησίας είναι ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο και βασίζεται, είναι δημοκρατία και αναγνωρίζει το Ισλάμ, την Ισλαμική θρησκεία ως την κυρίαρχη θρησκεία της Τινησίας. Υπάρχει αυτό λοιπόν. Ωστόσο, κάναμε μια ένθερμη θερμή συζήτηση με τον Άντα είναι ένα κόμμα το οποίο πρότεινε να υπάρξει και ένα προήμιο στο Σύνταγμα όπου να λέγεται, ε, όπου επιστρέφει σε μια συζήτηση που φαίνεται ξεπερασμένη ότι η θρησκεία είναι που να μιλά για τη θρησκεία ως κρατική θρησκεία και ε, που να μην περιγράφει απλώς ποια είναι η πρώτη θρησκεία στο, στην Τινησία. Το συνταγματικό δικαστήριο θα πρέπει να κρίνει ε, κατά πόσο ε, ε, το Σύνταγμα το Εθνικό εναρμονίζεται και με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Τινησία. Πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή αλλά καταλαβαίνετε ότι επί στη βάση αυτή θα αποφασιστεί το, το μέλλον όχι μόνο των γυναικών αλλά και της δημοκρατίας σε αυτήν την χώρη. Αυτό ήθελα να το θέσω γιατί είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Ε, το σήμα που θέλουμε να στείλουμε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο παρακολουθεί βήμα προς βήμα ε, το, την ψήφιση και την προετοιμασία του συντάγματος στην Τινησία. Ενδιαφέρεται πολύ το Συμβούλιο της Ευρώπης να λαμβάνει τις εκθέσεις που εμείς ε, συντάσσουμε και έχει και υπηρεσίες διασύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε. Τώρα ένας άλλος λόγος που είναι μικτός, λόγος αγωνίας και ελπίδας και που είναι και κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να μην το αποσιωπήσουμε, είναι ότι υπάρχουν λίγο δύο μέτρα και σταθμά του πιο τυπικού επίσημου επίπεδου και της κατάστασης που προσλαμβάνουν πολλές γυναίκες. Θυμάμαι την πρόοδο μιας σημαντικής ένωσης γυναικών επιχειρηματιών. Οι γυναίκες που ανησυχούν πάρα πολύ για την επιστροφή σε ένα παλιό καθεστώς αντιπροσωπεύουν το 40-45% των γυναικών και φοβούνται γιατί, γιατί υπάρχουν διαρκώς βιαιοπραγίες από φονταμενταλιστές, πολλοί από τους ε, φονταμενταλιστές έχουν επιστρέψει στην Τινησία από τις Ισλαμικές κοινότητες της Ευρώπης, να το σημειώσουμε αυτό, και ανησυχούν και πάρα πολύ οι γυναίκες αυτές γιατί υπάρχουν διαρκής πράξη εκφοβισμού, ε, καταστολής, βιαιότητας, με συγχωρείτε έτσι με συνεπέρνει το πάθος, ε, και μεγάλη πίεση στα μικρά κορίτσια και στους νέους ακόμα και στα πανεπιστήμια και για παράδειγμα σε αντάλλαγμα με σε αντάλλαγμα με κάποια υποτροφία για να σπουδάσουν, για να έχουν κάποιες περισσότερες ελευθερίες, πρέπει να φορέσουν τη μαντήλα. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Η οικονομία δεν πάει καλά. Λιγότερο 10% η βιομηχανική παραγωγή, λιγότερη προσέλευση τουριστών. Ε, υπάρχει η δυσαρέσκεια του πληθυσμού για τις οικονομικές δυσκολίες, η οποία είναι ένας παράγοντας που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, πιστεύω χρειάζονται τα δύο τρίτα της συντακτικής εθνοσυνέλευσης για την ψήφιση του συντάγματος. Εάν οι γυναίκες που είναι πολιτικά ενεργές συνενωθούν ε, να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ίσως να συντάξουν και ένα είδος οριζόντιας εκπροσώπησης, να το κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να επαφεθούμε μόνο σε ένα λαϊκό δημοψήφισμα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την κοινωνία. Δεν ξέρω εάν οι συνάδελφοι που είχαν έρθει μαζί μου ε, έχουν να προσθέσουν κάτι σε όλα αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τόσο αφοσιωμένους και παθιασμένους ε, βουλευτές. Θα αρχίσουμε τώρα τις ε, ψηφοφορίες, αλλά έχουμε την κυρία Γκάμπρελ, τον κύριο Ταραμπέλα. Δεν πρέπει να αργήσουμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία πρώτα από όλα που διοργάνωσε όλα τα ραντεβού και το ταξίδι της αντιπροσωπείας ε, να ε, ευχαριστήσω και τους αμφιτρίωνες. Ε, μας επιφύλαξαν καταπληκτική υποδοχή. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το πάθος και τον ενθουσιασμό της και τις βαθύτατες γνώσεις της, το οποίο θα αντανακλάται και στην έκθεσή της ίσως είμαστε μάρτυρες μια ε, ιστορική στιγμής, μιας ε, καμπής, ε, όπου όλα μπορούν να αλλάξουν. Μετά από αυτή την επίσκεψη μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τυνησίες. Μία σύγχρονη ανοιχτή, που όμως επικεντρώνεται γύρω στην πρωτεύουσα, και μία άλλη πολύ πιο κλειστή, όπου δεν υπερασπίζεται κανείς ανοιχτά τα δικαιώματα των γυναικών, εν είδη εφημισμού, αλλά Ε, και το κόμμα ΕΝΑΝΤΑ το οποίο ε, επικρατεί στις περισσότερες ε, περιοχές της χώρας. Θα έπρεπε να τονίσουμε ότι χρειάζεται να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος και το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πολλά περισσότερα πράγματα από μια διεξοδική έκθεση όπως αυτή της συναδέλφου Κώστα αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εγγράφουμε πάγια στην εμερήσια διάταξη το θέμα της Τινησίας ε, και του νέου συντάγματος. Εγώ θα επιμένω για τη σημασία του άρθρου 1 και 15 του προημίου που παραπέμπει στις διεθνείς συμβάσεις την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα και πρέπει εμείς να το παρακολουθούμε εκ του Σε Τέσσερα ζητήματα. Ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες των προστασία των κεκτημένων. Είδαμε σε ποιο βαθμό οι γυναίκες επί πού εφαρμόζουν τον προσωπικό κώδικα διοντολογίας. Χρειαζόμαστε τις απαιτούμενες ε, προϋποθέσεις, ούτως ώστε να συνεχίσει αυτός ο ακτιβισμός των γυναικών επιτόπου σε σχέση με τη συντακτική συνέλευση. Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για να αποφανθούν όλα τα πολιτικά κόμματα για τα δικαιώματα των γυναικών. Αφετέρου, οι αιρετοί εκπρόσωποι του λαού, οι γυναίκες πρέπει να εμπλακούν ενεργότερα οι ίδιες για την πρόθεση και προστασία των ε, δικαιωμάτων των γυναικών. Τρίτον, ε, ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία και η κρίση. Αυτό το ζήτημα των μικροπιστώσεων ε, και όλη η συζήτηση που έγινε γι' αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό το 20% που αναφερθήκατε μου φαίνεται πολύ περίεργο και είναι επικίνδυνο αυτό για την υπερχρέωση. Δηλαδή είδαμε πολλές περιπτώσεις γυναικών που είχαν μία πρώτη μικροπίστωση, δεύτερη, τρίτη, οπότε δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι είναι καλή αυτή η ιδέα. Σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών χρειάζεται καλή ε, επικοινωνία ούτω ώστε να προωθήσουμε μία πιο ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία οικονομική ζωή και στις ανώτερες θέσεις επιχειρήσεις. Τώρα ως προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές φωνές κατά της δράσης της Ένωσης για το ρόλο της στην Τινησία όμως έχει διπλασιάσει τα κονδύλια που χορηγεί στην Τινησία ε, βεβαίως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με ε, την θέση που παίρνουμε για δύο βασικά ζητήματα, για τη γεωργία και τη μετανάστευση ή γενικότερα για όλα τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Ε, να είμαστε σε ε, γρήγορες λοιπόν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για αυτά τα δύο κεντρικά ζητήματα ε, και να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτό το θέμα της Τινησίας. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια, ευχαριστώ τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο γιατί καταδεικνύουμε έτσι το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τη χώρα αυτή και δείχνουμε ότι δεν πρόκειται για μια απλή επίσκεψη ε, πρωτοκόλου ε, τυπική, αλλά ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τις εξελίξεις σε αυτή την χώρα. Σας ευχαριστούμε και τώρα σας ακούσουμε τον κύριο Ταραμπέλα για μια σύντομη παρουσίαση της επίσκεψης εκεί. Έχετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ τη Σίλβια Κώστα και για την έκθεσή της, αλλά και για το λόγο της που δεν θα το κρύψω. με εντυπωσίασε. Στην ναι, Ισία μιλήσαμε για αραβική ανοίξη, αλλά πρόκειται για φθινόπωρο, ε, αραβικό φθινόπωρο ή αραβικό χειμώνα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, μέσα σε αυτή την έκθεση λέμε δεν πρέπει να στιγματίζουμε κανέναν. Ε, λοιπόν όχι. Γιατί να μην καταγγείλουμε ε, την, τον εκτροχιασμό που παρατηρείται στην την Όντως να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις προσπάθειες τους αλλά ε, ε, ε, αυτό που ε, μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση είναι η Νάρτα που ανεβαίνει στην εξουσία που θεωρείται ότι είναι ε, το συμπλήρωμα του, το αντρικού φύλου. Δεύτερον, ε, την έχουν εκθιάσει και έχει ουσιαστικά αναδειχθεί σε σύμβολο της χώρας ε, ενώ πρόκειται για μια απλή δρομέα ε, και σε άλλες χώρες δεν τις έχουν επιφυλάξει την ε, ίδια μεταχείριση. Θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτήν την οπισθοχώρηση της Τινησίας. Αντικαθιστά μια δικτατορία με μια θρησκευτική δικτατορία και αυτό ισχύει και για άλλες χώρες και γι' αυτό σας μιλάω για αραβική, αραβικό φθινόπορο. ελπίζω ότι με την έκθεση της κυρίας Κώστα θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Δεν ξέρουμε πώς καταρτιστεί τελικά και η έκθεση πρωτοβουλία πρωτοβουλία ή κάποιο άλλο έγγραφο, αλλά πάντως ε, θα πρέπει να μιλήσουμε ε, ειλικρινά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ξύλινη γλώσσα, γιατί δεν είμαστε διπλωμάτες, είμαστε πολιτικοί και είναι δυσάρεστο και μα θορύβει αυτά ε, αυτό που συμβαίνει στην Τινησία και θα πρέπει να εκδηλώσουμε την διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας προς τις τελευταίες εξελίξεις. Σας Ευχαριστούμε και ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα μεταγενέστερα. Ε, υπήρχε και η κυρία Γκαμπριέλ από το ΕΛΚΑ και η κυρία Νικόλ Νίλσεν από τους Περασίνους, πέρα από την εισηγήτρια και από μένα τον ίδιο στην αποστολή. Το ξέχασα αυτό προηγουμένως, δεν σας το είπα. Ας περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. Okay, we will then start the voting Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Η πρώτη είναι η εξάλληψη των συνδεωμένων με το φύλλο στερεοτύπων στην Ένωση. Η κυρία Καρτίκα Λιωτάρ που είναι η συγγήτρια θέλει να μιλήσει τώρα. Ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πολλές ήταν μια προσθήκη και μια βελτίωση της έκθεσης. Ευχαριστώ και πάλι όλους και έχουμε καλά αποτελέσματα από την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε να ψηφίσουμε, ανακοινώνω ότι είναι μόκρα ο κατάλογος ε, της ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε και unblock μερικές φορές, αλλά θα σας ζητήσω να συμφωνήσετε από πριν. Και αν διαφωνεί κάποιος δεν θα το κάνουμε. Αλλά θα κοιτάξω να δουλέψουμε ψηφίζοντας ε, unblock και υπολογίζω στην βοήθειά σας για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πρώτη τροπολογία έχει αποσυρθεί η πρώτη. Ε, πάμε στην 81, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Ε, η 81, η 83 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 85 κατά πίπτη, πάμε στη συμβιβαστική ε, ε κατά αποχές δεκτή. Μετά πάμε στην τροπολογία 90, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 95, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 96-97 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 98 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία τώρα The vote is closed. Πέρας. Δεκτή. 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 100 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε απερίφθη με διαφορά δύο ψήφων, η 101 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Και τώρα είναι δυνατόν να πάμε από την 102 μέχρι την επόμενη σελίδα την 146. Όχι. χωρίς ε, μικρόφωνο οι παρεμβάσεις. Δηλαδή να τις ψηφίσουμε μία προς μία. Καλώς. 102 με 122. Όχι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Μία, μία προς μία θα τις ψηφίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Η 102 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 και 107 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 108 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 110 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 111 και 112 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να ελέγξουμε την 111 και την 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται με διαφορά μιας ψήφου. 113-116 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 114 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ελέγχουμε την 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 115-118. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Οι 117 και 119 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 122 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Είναι δυνατόν να πάρουμε τώρα τίποτα unblock. Όχι, όχι. Εντάξει, απλώς ρώτησα. Πάμε στην 123. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή 130 υπέρ κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 και 135 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή 139 υπέρ κατά αποχές δεκτή 140 υπέρ κατά Αποχές δεκτή. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 145 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε έλεγχος. Ελέγχουμε την 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 145. Δεκτό, δεκτή. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 147 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε την 147. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει ένας. Πέρας. Απερίφθη με διαφορά μιας ψήφου. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρα πάμε στο 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 156 και 157 ταυτόσημες. Ε, και οι 158. Και οι τρει υπέρ, ποιο είναι και των τριών, κατά, αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 163. Είναι δυνατό να πάμε από την 163 μέχρι την 185. Ναι. Χωρίς σε μικρόφωνο Εκατόν 163-165 Ταυτόση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 164 άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Πέρας. Απερίφθη. Απερίφθη. 10 προς 10. 10 υπέρ, 10 κατά. Πάμε στην 166. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 167-168 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 169 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 170 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 171 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή 181 και 182 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 183 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 184 και 86 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 185 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Είναι δυνατόν την 1 ε, με 10 τροπολογίες να την πάρουμε, να τις πάρουμε όλες μαζί. Α, μάλιστα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία, τη συμβιβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική 2. Όχι, προχώρησα πολύ. Όχι, ψηφίζουμε την τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Η 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Α, όχι, όχι, καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική 2 τώρα. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και πάμε τώρα στην 21 και 22 που είναι ταυτόσιμες. 24, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 22, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 και 25 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές 27 υπέρ όχι όχι την 26 ήθελα να πω ε, υπέρ της 26 κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή πάμε στη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές Για μισό λεπτό θα ελέγξουμε για να είμαστε βέβαιοι. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 3. Πέρας. Δεκτή με μια ψήφο διαφορά. Τώρα. Πάμε στην 34. Είναι δυνατόν να πάμε μέχρι τις 40 να ψηφίσουμε όλες. Όχι. Καλά. 34 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να ελέγξουμε την 36. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 36. Πέρας. Απερίφθη. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 39. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 και 56 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα, ξανά θα επιχειρήσω. με 51. 43 να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 45 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 46 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 50 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 53 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 είναι μια προφορική τροπολογία έχετε διαφωνία ψηφίζουμε την 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 71 και θα προσπαθήσω και πάλι από την 71 μέχρι την 77. Όχι. Πάμε στην 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 74. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές. Δεκτή. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 76 και 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή και πάμε να ψηφίσουμε όλο το ψήφισμα, το τελικό. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά θα το ψηφίσουμε. Λείπει μία ψήφος. Πέρας. Και εγκρίνεται. Δεν λειτουργήσε το δικό σας, προσθέτουμε μία θετική ψήφο. Σαφώς εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια. Okay, we then go to the next. Θα περάσουμε ε, στον επόμενο κατάλογο ψηφοφοριών ε, σε σχέση με την ενσωμάτωση των μεταναστών και τις επιπτώσεις αυτού στην αγορά εργασία και την εξωτερική διάσταση της συντονισμού για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η συγκίτρια θα ήθελε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ επίσης για τις ε, τροπολογίες που υποβάλατε. Χάρη σε αυτές είναι σαφέστερο και περιεκτικότερο το έγγραφο. Η Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολείται με το ζήτημα συχνά και εγώ μετέχω σε αυτή την Επιτροπή και ε, συχνά συναντούμε με μετανάστριες γυναίκες και πιστεύω ότι χάρη στην έκθεση θα μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική ε, συνεισφορά για την ενσωμάτωση αυτών των γυναικών σας ευχαριστούμε η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ Έλεος δείξτε, διότι η πρώτη παρέμβαση είναι που κάνω και η πρώτη τροπολογία σε αυτή την επιτροπή. Πρόκειται για την υπαριθμό 7. Λέει στον κατάλογο ότι αν η τροπολογία 1, η 5 και 6 εγκριθούν, καταπίπτει η τροπολογία 7. Εγώ θεωρώ ότι δεν καλύπτεται από τι συμβαστικέ τροπολογίε η δική μου, γιατί μιλάει για τι μετανάστε συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μετακινούνται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και υφίσταται βία κτλ. Βλέπετε είναι διαφορετικό. Ήθελα να τονίσω με την τροπολογία ότι πολλέ ε, γυναίκε πολίτε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ουγγαρία παραδείγματο χάρη ε, που μετικούν στη Δυτική Ευρώπη για να εργαστούν σε άλλε χώρε, υφίστανται διακριτική μεταχείριση, πέφτουν θύματα εμπορία ανθρώπων και πλήττονται από διάφορα φαινόμενα που εξετάζουμε εδώ στην Επιτροπή μα. Δεν καλύπτεται ω εκ τούτου η τροπολογία μου από τι συμβαστικέ τροπολογίε και θα συνιστούσε χρήσιμη προσθήκη, ε, δηλαδή ε, η ουσία της τροπολογία μου είναι να καλύψουμε και τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωση που μετακινούνται στο εσωτερικό τη Ένωση και να τη συνδυάσουμε με τη σχετική συμβαστική τροπολογία και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Okay, you put me in a quite tricky... Μάλιστα, με θέσατε σε μία λεπτή θέση ε, και Καταλαβαίνω γιατί γύρατε το ζήτημα, όμως όταν καταρτίζει κάποιος κατάλογο ψηφοφορίας ε, θα πρέπει, πρωτού καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος, να ξέρουμε τι πρόσημο έχει. Ε, οπότε ε, έτσι ξέρουν όλοι πώς θα κινηθούν στην ψηφοφορία. Ενδέχεται, από ό,τι καταλαβαίνω, να ψηφίσουμε χωριστά την τροπολογία σας Καταπίπτει όμως αν εγκριθούν άλλες τροπολογίες, αυτά που σας έλεγα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη χρονική στιγμή να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, προτού καταλήξουμε στον τελικό κατάλογο ψηφοφορία, παρακαλώ να παρέμβετε σε μια, ε, για ένα επόμενο θέμα, διότι μόνο τότε μπορούμε να ελέγξουμε αν είναι δυνατόν κτλ. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά θα την ψηφίσουμε την τροπολογία σας σε χωριστή ψηφοφορία, αλλά δεν θα την εντάξουμε σε κάποια άλλη για να ξέρουν όλοι πώς θα κινηθούν. Οπότε θα ψηφιστεί η τροπολογία σας, μην ανησυχείτε, παρόλα αυτά. Αρχίζουμε. 14 υπέρ παρακαλώ. Κάτα. ηχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε απευθείας συμβαστική υπαριθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Αυτό σημαίνει ότι περνούμε στην ε, τροπολογία 28 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 31 είναι κατά τμήματα ψηφοφορία. Αρχίζουμε με το πρώτο, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα για την τροπολογία 32 που επίσης είναι κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 τώρα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα θα ήταν να το εξακριβώσουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Λείπουν τρεις, δύο, ωραία, πέρας ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ξεκάθαρα. Η 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 είναι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 56 τώρα. Θα μπορούσαμε από τη, ομού να ψηφίσουμε από την 56 έως την 63. 62 θέλετε. Οκ, 62. 56 έως 62 ομού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε στην 9 Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινό όλε τι υπολοιπόμενε τροπολογίε. Ωραία. Από την 9 στη 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Ε, εγκρίθηκαν. Ε, ψηφοφορία για το σύνολο. Διακόπτη ένα μέλο επιτροπή εκτό μικροφώνου. Ζητά συγγνώμη ο πρόεδρο. Ε, είχα βυθιστεί μέσα στο κατάλογο ψηφοφορίας και ξεχάστηκα. Πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 7, όπως ε, υποσχέθηκα προηγουμένως. Όχι, η κυρία Μορβάη, δεν θυμάστε, είπε ότι δεν συμφωνεί, ότι καταπίπτει η τροπολογία. Μίλησα με τη γραμμάτια και θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστή ψηφοφορία αυτή η τροπολογία. Η δική μου θέση είναι ότι καταπίπτει, αλλά τη προσφέρω την ευκαιρία παρόλα αυτά να ψηφιστεί, να γίνει ψηφοφορία για την τροπολογία τη. Θα την ψηφίσουμε ούτω ή άλλω η τροπολογία 7 για να έχετε την ευκαιρία σα, ε, κυρία Μορβάη. Ποιοι είναι υπέρ τη τροπολογία 7 παρακαλώ. Κατά τώρα. Αποχέ Απερίφθη. Συμφωνώ μαζί σας ότι έτσι έχουμε τα πράγματα, αλλά συζητήσαμε προηγουμένως και ήθελα να τη δώσω την ευκαιρία να γίνει ψηφοφορία για τροπολογία. Δεν είναι αρμοδέτα του Προέδρου ούτως ή άλλως Επιτροπής να το αποφασίζει από τη 19 στην 30 υπέρ κατά. Και αποχές. Εγκρίθηκαν. Ναι, ναι, το ξανά έκανα γιατί δεν ήξερα αν ε, θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 7. Τέλος πάντων, ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο ε, της έκθεσης, ε, ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφο. Όχι, εντάξει, ωραία, πέρας. Ναι, εγκρίθηκε με 12 ψήφους προς 8. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, και εσύ, έλα, να χασμοριθώ Προστασία της δημόσιας υγείας. Ελπίζω να μπορέσουμε αυτό να το ψηφίσουμε unblock. Εντάξει, να το ψηφίσω, να το προτείνω έτσι. Κοιτάζω και το ΕΛΚ. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. We then go to the final... Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Το σχέδιο προφορικής ερώτησης ε, για την ε, ε, βία κατά των γυναικών. we Πριν από την προθεσμία λάβαμε δύο προτάσεις τροποποίησης του σχεδίου κειμένου. Τώρα έχουμε την ενοποιημένη εκδοχή, έχουμε συνδυάσει τα δύο δηλαδή αν έχω, αν πληροφορηθεί σωστά, εχθές υπήρξε μία υπόδειξη από τους σοσιαλδημοκράτες στην στο ενοποιημένο κείμενο μας ζήτησαν αν μπορούμε κάτω-κάτω εκεί που λέει ε, στην ερώτηση δύο, η επόμενη πρόταση, ένα πρώτο βήμα προς κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, το βλέπετε? Το πρώτο βήμα, ένα πρώτο βήμα προς κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θα το θεωρήσουμε αυτό ως προφορική πρόταση τροποποίησης. Ε, την αλλαγή αυτών των λέξεων που μόλις σας διάβασα. Με παρακολουθείτε? Συμφωνείτε να έχουμε αυτή την τροποποίηση? Αν λοιπόν ε, δεν θέλω τώρα να έχουμε διαφορετικές προτάσεις θέλω να έχουμε μία πρόταση, την το ενοποιημένο κείμενο με τον συνδυασμό αυτών. Κύριε Μπάουερ, συγγνώμη, το ξέρω ότι είναι αργά για να θέτει κανείς ερωτήσεις, αλλά ε, μου φαίνεται πως είναι κρίμα να μην συμπεριλάβουμε και την η υπόσχεση της Επιτροπής. Όπως θα θυμάστε, η κυρία Ρέντινγκ υποσχέθηκε για αυτήν την πρόταση ε, καταπολέμησης της βίας των γυναικών. Πρότεινε να υπάρξει ένας κανονισμός πάνω σε αυτό. Ε, ήταν μια σαφής υπόσχεση από την πλευρά της ε, στις αρχές. Ε, γιατί να το αφήσουμε απ' έξω. Επίσης, κάτι άλλο που λείπει είναι ε, μια έκκληση για ολοκληρωμένες πολιτικές. Ε, ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική δεν λαμβάνει ιδιαίτερος υπόψη της την πολύ υψηλή συχνότητα της διάπραξης ε, βιαιοτήτων κατά των γυναικών σε πολλές νότιες αφρικανικές χώρες ή χώρες της Καραϊβικής ή στην Κίνα. Κάτι που θα το, θα, για το οποίο θα ενημερωθούμε και με μία έκθεση ως ούπο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο μεγάλα θέματα δεν θα έπρεπε να λείπουν. Ε, το ξέρω όμως ότι ε, έρχομαι πολύ αργά με αυτές τις προτάσεις. Το συνειδητοποιώ. Ναι. Ε, είναι λίγο προβληματικό να γυρετε τα θέματα αυτά τώρα αλλά πάντοτε έχετε τη δυνατότητα να το θέσετε ως προφορική τροπολογία. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την έγγραφη διαδικασία, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τους υπόλοιπους, για τα άλλα μέλη της Επιτροπής, να γνωρίζουν επαρκώς ε, πώς θα διατυπωθούν ακριβώς οι προτάσεις σας. Δεν ξέρω ε, αν έχετε την ευκαιρία να γράψετε μέσα σε ένα λεπτό μια προφορική τροπολογία. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, θα έπρεπε να το έχω ελέγξει. Εάν ήταν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ή αν ήταν πρόβλημα του Συμφώνου για τα φύλλα που ανακοίνωσε η κυρία Ρέντινγκ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ε, θυμάμαι ακριβώ μόνο το περιεχόμενο τη υπόσχεση, αλλά όχι πότε δόθηκε αυτή η επευκαιρία ποιου προγράμματο. Η κυρία Κονέλης. Ίσως μπορεί η Επιτροπή να ψηφίσει, να δώσει εντολή στου συντονιστέ να συντάξουν μια τέτοια επιστολή, αν όλοι πιστεύουμε ότι η κυρία Μπάουερ έχει δίκιο. Ε, Πρόεδρο, κύριο Γκούσταυσον. Ναι, πραγματικά μπορεί να γίνει γιατί έχουμε συνάντηση των συντονιστών. Οπότε μπορούμε να αποφασίσουμε ότι υιοθετούμε την ενοποιημένη, το ενοποιημένο κείμενο και οι συντονιστές μπορούν να εισαγάγουν κάποιες τροποποιήσεις με βάση την πρόταση της κυρίας Μπάουερ ή κάτι τέτοιο. Κυρία Κιβέτη, κατά την γνώμη μου φυσικά έχει δίκιο η κυρία Μπάουερ, αλλά ταυτόχρονα όταν λέμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να έχει την ολοκληρωμένη πολιτική και τα νομικά εργαλεία. Νομίζω ότι εδώ συμπεριλαμβάνεται η πρωτοβουλία και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι ο τρόπος που έχει γίνει η διατύπωση στο έγγραφο που έχουμε μπροστά μας περιλαμβάνει αυτή την ολοκληρωμένη πολιτική και την υπόσχεση της κυρίας Ρέντινγκ. Ε, ήθελα απλώς να το θέσω. Ναι. Ε, εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο προφορικών ερωτήσεων, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, αλλά μπορούμε πράγματι να ρωτήσουμε τους συντονιστές να επιφέρουν κάποια τροποποίηση, εάν θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η κυρία Τσούμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε όσο έχει το κείμενο. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που όλοι θεωρούν ότι είναι η ολοκληρωμένη στρατηγική της καταπολέμησης της βίας, ε, έχει διάφορα είδη βίας ε, κατά των γυναικών και έχουμε και το θέμα του ακροτηριασμού των ε, γεννητικών οργάνων των γυναικών που υπονοείται στο κείμενο. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε συγκεκριμένα κατά τη γνώμη μου στα διάφορα μεμονωμένα είδη βίας κατά των γυναικών, ε, όμως ε, καλό θα ήταν να διευρύνουμε τη συζήτηση στη συνεδρία των συντονιστών. Εγώ θα ήμουν υπέρ. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος, θα ήθελα να είμαι σαφής. Ε, εάν δεν υπάρχουν στάσεις ε, κατά αυτής τη πρόταση, τότε σημαίνει ότι καταπίπτει γιατί ε, επέχει θέση προφορικής τροπολογίας και ω εκ τούτου δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία. Όμως, ε, αν λάβουμε μια απόφαση βάσει της οποία θα δεχθούμε την ολοκληρωμένη μορφή, ε, τότε αν κρίνουν σκόπιμο οι συντονιστέ να τροποποιήσουν το κείμενο δυνάμει της πρότασης αυτής, τότε είναι επιλογή τους, αλλά επαφείται στην κρίση των συντονιστών ε, να διαπιστώσουν αν ε, χρειάζεται αλλαγές το κείμενο ή όχι. Ακόμη και ένα να προβάλλει ένσταση καταπίπτει, γιατί, ξαναλέω, επέχει θέση προφορικής τροπολογίας. Σας κοιτάζω τώρα για να μου πείτε. Oh. Compromise proposal, ε, could that be a good way to deal with That... Ε, μήπως να τα αφήσουμε στους συντονιστές, μήπως αυτός θα είναι ένας ε, καλύτερος τρόπος να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Δεν θα εφαρμόσουμε τη θέση τη κυρίας Μπάουερ, θα το αφήσουμε στους ε, συντονιστές. Δηλαδή σε μια σύσκεψη μικρότερης, πιο περιορισμένη σύνθεση καλό θα ήταν να συζητηθεί το θέμα αυτό, ενώ συμφωνείτε όλοι μαζί μου. Πολύ ωραία. Α, η κυρία Κώστα. Ε, να πω μόνο ότι θεωρώ αν, αν όλοι επιθυμούμε τον ίδιο σκοπό να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες βίας, ίσως οι συντονιστές να μπορέσουν να εισαγάγουν κάποια τροποποίηση, αλλά να λένε any kind of violence, κάθε τύπο βίας. Δηλαδή να υπογραμμίσουμε ότι δεν εξαιρείται κανένας τύπος βίας, καμία μορφή βίας. So once again, because I want really be... Και πάλι γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο το ζήτημα για να ξέρουν όλοι για ποιο θέμα θα τοποθετηθούμε. πρώτο προτείνω να εγκρίνουμε την ολοκληρωμένη εκδοχή, δηλαδή συμπεριλαμβανομένες τροπολογία που προέρχεται του σοσιαλιστές και δημοκράτες και κατά δεύτερο λόγο να αφήσουμε στην κρίση των συντονιστών την απόφαση αν χρειάζεται αλλαγή το κείμενο σύμφωνα με την πρόταση της κυρίας Μπάουερ. Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αυτό ω Επιτροπή. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά τώρα. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση αυτή. And uh, the final, uh, Ορίστε κύριε Μορβέ, ζητώ συγγνώμη πριν κλείσετε τη σημερινή συνεδρίαση να καταγραφεί τα πρακτικά γιατί αναμεταδίδεται και η συνεδρίαση. Είναι μαύρη η σημερινή ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη, γιατί η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής αποφάσισε σήμερα ότι οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γυναίκες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, που είναι υποχρεωμένες λόγω των παγκοσμίων ανισοτήτων να μετικήσουν σε πλουσιότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δικαιούνται την ίδια νομική και άλλη προστασία όπως οι πίκοοι, οι από τρίτες χώρες, ε, από την Αφρικανική Ήπειρο παραδείγματο χάρη έσχος και κυρίως ε, για τα μέλη της Επιτροπές που προέρχονται από αυτές τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης γνωρίζουν πως οι αδελφές και συμπατριώτητές τους υποφέρουν όταν δουλεύουν ε, και υφίστανται κατάφορη εκμετάλλευση, παραβίαση των δικαιωμάτων τους όταν εργάζονται ως οικιακή βοηθή, παραδείγματος χάρη, ντροπή και έσχος που απέρριψαν την τροπολογία μου, γιατί χάρη σε αυτήν θα εξασφαλίζαμε ισότιμη προστασία όπως και για τις, τους πολίτες τρίτων χωρών. Όλοι ήξεραν ε, για ποιο λόγο υπέβαλα την τροπολογία. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σε επαναφέρω στην τάξη για δύο λόγους. Μα δεν είστε πρόεδρος, πώς θα με επαναφέρετε μετά στην τάξη. Κύριε Μορβάη, Συγγνώμη, αλλά για τα πρακτικά, γιατί όλα λέμε για την ελευθερία τη έκφραση και είναι δικαίωμά μου βάσει αυτού του δικαιωμάτου και ε, ε, οι εκλογεί δικαιούνται να ξέρουν ότι είμαστε εδώ και έχουμε παχυλότατου μισθού και αντί να εξασφαλίσουμε προστασία για αυτέ τι γυναίκε, καταψηφίζουμε την πρόταση βάσει τη οποία θα εξασφαλιζόταν ισότιμη νομική προστασία κατά τη εκμετάλλευση αυτών των γυναικών έσχο. Ήθελα να καταγραφεί. Πρόεδρος, θα δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία Μπάουερ δεν μ' αρέσει ακριβώς να μιλάμε για αυτόν τον τρόπο με αυτά που συμβαίνουν. Ζητώ συγγνώμη, ψηφίσαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε ε, πράγματα για εσωκομματική κατανάλωση. Έτσι εντάξει, ωραία, καταγράφηκε στα πρακτικά αυτό που είπατε, τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή κύριε Μπάουερ. Θα μιλήσω ουγγρικά για να μην ε, παρανοηθώ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ε, και ξέρετε τι έγινε και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, εχθές ε, σχετικά με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αυτή η έκθεση φέρει επί του θέματος της μετανάστευσης από τις τρίτες χώρες και το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κατά πόσο η τα κινούμενοι εργαζόμενοι καλύπτονται από τα συστήματα της κοινωνικής ε, ασφάλισης. Ήταν αυτή, ε, ε, έγιναν όλα οι καλών προθέσεων. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το τόνο της κυρίας Μορβάη ε, κοίταξτε, λέει η κυρία Κορνέλη, ε, ναι, πρέπει να την επαναφέρουμε σε τάξη την ε, κυρία Μορβάη, διότι δεν επιτρέπουμε σχόλια και παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει κανείς και κυρίως όχι με αυτό το ύφος. Ε, οπότε εκτροχιάζεται η κυρία Μορβάη ε, και Μιλάει για διαφορετικέ σκοπιμότητες για τον τρόπο που ψηφίσαμε. Εγώ καταψήφισα την τροπολογία διότι ομαδοποιείται ε, τις ε, μετανάστες γυναίκες από τρίτες χώρες και τις ταξινομείται στην ίδια κατηγορία με τις ε, γυναίκες που εσωτερικά μετακινούνται στο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάγονται όμως σε λίγα διαφορετικά καθεστώτα και δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις δύο κατηγορίες και μην τεκμέρετε κυρία Μορβάη ποιε είναι οι σκοπιμότητές μας για το όταν ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Λούλη. Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτήν την ε, τροπολογία διότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ε, <laughs> πρέπει να ξέρω ότι όταν μετικό από τη μία χώρα στην άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας. Ε, από την ΕΚΑΧ ε, έχει κατοχυρωθεί αυτό είναι, τι να σας πω, καμία σχέση με το θέμα. Είμαστε εκτός θέματος. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ε, συγκεχημένα όλα τα πράγματα στο μυαλό των ε, ε, νεόφερτων σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια τροπολογία που είναι εκτός θέματος, αλλά αντάλλων θα έλεγα. Θα τα πω στα σου ειδικά γιατί είναι σημαντικό να περάσει το μήνυμα. Κυρία Μωραή. Ακριβώς ε, τέτοιου είδους καταστάσει θέλω να αποφεύγω στην Επιτροπή. Δηλαδή μετά το πέρασε των ψηφοφοριών αρχίζει συζήτηση για την ερμηνεία της ψήφου του καθενός. Δεν γίνονται αυτό ορισμένε φορές και εγώ κρίνω ότι είναι ε, σφαλμένη θέση ε, της Επιτροπής μας. Αλλά δεν είναι η σωστή θέση και χρονική στιγμή για να συζητούμε για την έκβαση της ψηφοφορία εδώ. Εκτός μπορείτε, γιατί είναι θέμα πολιτικής και υπάρχουν και ανακοινοθέντα τύπου κτλ. Αλλά δεν γίνεται μετά από κάθε ψηφοφορία να γίνεται αυτό. Εσείς καλά κάνατε και ζητήσατε το λόγο και κάθε φορά θα σας τον δίνω. Όμως δεν γίνεται να συζητάμε ε, το πώς ψήφισε ο καθένας ε, μετά από κάθε ψηφοφορία. Δηλαδή αυτό θα ε, ήταν μια τέρμονη διαδικασία. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο και ούτως ή στη πολιτική δεν κάνουμε μέσα στην Επιτροπή, εκτός αιθούση τι κάνουμε. Ε, παρακαλώ, θα σα ξαναδώσω το λόγο παρόλα αυτά, αλλά πολύ σύντομα να είστε. Yes, I, I think you shouldn't uh, be so worried about... Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τη δημοκρατική συζήτηση εν κενό. Ε, Ευρώπη και δημοκρατία σημαίνει οι πολίτες της Ευρώπης να αποφασίζουν οι ίδιοι τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφτιλίζει τη χώρα μου, την Ουγγαρία, εδώ και χρόνια ότι δεν είμαστε παρκώς δημοκρατικοί. Εσεί πώ είστε τόσο κακοί και ανέχεστε μια τέτοια συζήτηση. Έτσι ακριβώ πρέπει να λειτουργεί η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που τώρα έχουν διασαφινιστεί οι θέσει και θα εξασφαλίσω ότι στο διαδίκτυο θα διατεθεί η συζήτηση αυτή έτσι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε να την παρακολουθήσουν και να λάβουν μόνοι του τι αποφάσει του. Συγγνώμη, πρέπει να λήξει αυτή η συζήτηση και μετά τη λήξη της συζήτησης σα κάνουμε όλη πολιτική εκτός ε, αιθούσης, αλλά όχι μετά την διαδικασία της ε, ψηφοφορίας, ε, γιατί δεν γίνεται να κατασπαταλούμε έτσι το χρόνο της Επιτροπής κάθε φορά που ψηφίζουμε και κάθε φορά που κάποιος καταψήφισε, κάθε αρχίζει τέτοια συζήτηση. Εγώ αυτό εννοώ. Δεν σας αρνούμε το λόγο, σας δίνω το λόγο, δεν ε, παραβιάζω την ελευθερία έκφρασή σας, απλώς είναι μια σύσταση από πλευρά μου. Λοιπόν, επόμενη συνεδρία, όχι, ε, σημείο 11 συνεδρία των συντονιστών θα γίνει ευθύ αμέσω. Πάντω, η επόμενη συνεδρία θα γίνει 17 και 18 Δεκεμβρίου στις 10 17 ε, Δεκεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και στις 18 από τις 9 ως τις 12.30 τη λήξη τη συνεδρίαση ε, και σε δύο λεπτά περίπου θα ε, αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών παρακαλώ.